Τροπής είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την κατάσταση στην νοτιοανατολική Τουρκία και ο πρώτος ομιλητής ε, που εκπροσωπεί την κυρία Μογκερίνη είναι ο Επίτροπος ο Γιωχάνης Αν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα σήμερα η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας ε, στην νοτιοανατολική Τουρκία είναι πολύ ανησυχητική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες της για την κατάσταση και το, στις 22 Σεπτεμβρίου και τον Ιανουάριο πιο προσφάτως και παρακολουθούμε την κατάσταση στενά. Τα προβλήματα και στις ε, δύο πλευρές έχουν επίσης επιδεινωθεί από την ε, τρέχουσα κρίση και την απειλή από το Ισλαμικό κράτος όπως έδειξε και η τελευταία επίθεση του Κωνσταντινούπολη στις 12 Ιανουαρίου και οι επιθέσεις πέρσι στην ε, Άγκυρα και αλλού. Όμως η Μέση Ανατολή και η σταθερότητα είναι σημαντική όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή. Πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε τον πολιτικό χώρο που δημιουργήσαμε με κόπο για να ξεκινήσει μια μετάβαση στην Συρία. Η μόνη δυνατή και αποτελεσματική αντίδραση είναι να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις που έχουμε στην περιοχή μας με ενιαίο τρόπο. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το Ισλαμικό κράτος επί τόπου. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην διαλυθεί η κουρδική ειρηνευτική διαδικασία και να μην ε, πυροδοτηθούν νέες εντάσεις. Σε κάθε μας επαφή με την Τουρκία παροτρύνουμε όλα τα μέρη να εγγυηθούν το κράτος δικαίου και, το κράτος δικαίου και ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στην ειρηνευτική διαδικασία. Ο διάλογος ε, υψηλού επίπεδου στις 25 Ιανουαρίου θα είναι άλλη μια ευκαιρία να θίξουμε αυτά τα ζητήματα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε εδώ και μια γενιά για να λυθεί μια σύγκρουση η οποία έχει κοστίσει πάρα πολλέ ζωέ επίση ήταν σαφέ ε, πως το ΠΚΚ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά της Τουρκίας να συνεχίσει, να σταματήσει να ανακηρύσει αυτονομία στις ε, περιοχές ε, τι νοτιοανατολικές και ο διάλογο είναι ο μόνος δρόμο που υπάρχει. Θα συνεχίσουμε να διαβαίνουμε την Τουρκία πω η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ στα σοβαρά την απειλή του ΠΚΚ και πως τα κράτη-μέλη επίσης έχουν δράσει στεναρά κατά του ΠΚΚ. Το ΠΚΚ είναι μια οργάνωση που βρίσκεται σε κατάλογο κυρώσεων από το 2002. Το Συμβούλιο ομοφόνος ενέκρινε αυτή την απόφαση το Μάρτιο του 2015 και έτσι θα παραμείνει η κατάσταση για το προσεχές μέλλον. Όμως παρά το ότι αναγνωρίζουμε το θεμητό δικαίωμα της αυτοάμυνας στην Τουρκία κατά του ΠΚΚ τονίσαμε επίσης και θα συνεχίσουμε να τονίζουμε στον διάλογο με τις τουρκικές αρχές πως τα μέτρα που λαμβάνουν κατά του ΠΚΚ πρέπει να είναι αναλογικά, στοχευμένα και να μην θέτουν σε κίνδυνο το δημοκρατικό πολιτικό διάλογο. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν τώρα οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Νοτιοανατολική Τουρκία που ε, περιλαμβάνουν απαγόρευση κυκλοφορίας οδηγούν ε, σε δυσκολία στην παροχή βασικών υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες υγείας ε, και οι επικοινωνίες και οι συγκοινωνίες. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συμμορφώνονται με τις διεθνείς διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάποια από αυτά τα ζητήματα υπάρχουν επί δεκαετίες και θα απαιτηθεί θάρρος από όλες τις πλευρές για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν θα συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση για μεταρρυθμίσεις στον τομέα του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της θρησκείας και βέβαια αναμένω και την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στους ομιλητές ε, εξ ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρώτα η κυρία Ζόμερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Τι υπάρχει στην Τεντολκησία. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία στον Διαμπακύρ. Οι ε, ένοπλε δυνάμει τη Τουρκία επιτίθενται κατά το άμοχο πληθυσμού. Πολλέ ε, γυναίκε και παιδιά, νεκροί ή νεκροί, είναι απλά πεταμένοι στου δρόμου και δεν μπορούν να θαυτούν γιατί οτιδήποτε κινείται το πυροβολούν. είναι η κατάσταση σε 17 κουρδικές πόλεις. Μοιάζει με πολιορκία. Υπάρχουν ε, προβλήματα στην τροφοδοσία, όχι μόνο με το ρεύμα και το διαδίκτυο, δεν έχουν καν τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατάσταση είναι απάνθρωπη. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πόλεις και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν πληγεί, 250.000 βρίσκονται σε φυγή. Από ό,τι φαίνεται, οι δηλώνουν υποτίθεται ότι είναι ο αγώνας κατά του ΠΚΚ. Δεν είναι έτσι. Είναι ο αγώνας κατά των Κούρδων στην πλάτη του άμαχου πληθυσμού. Ε, η περιοχή αυτή έχει γίνει εμπόλεμη περιοχή και δεν επιτρέπεται λοιπόν να ε, συμπεριφερόμεθα με μετριοπαθή τρόπο. Δεν είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη, εμείς ε, λόγω του προσφυγικού να κλείνουμε τα μάτια και μόνο αυτό, αλλά να επιβραβεύουμε την τουρκική κυβέρνηση και με το άνοιγμα νέων κεφαλαίων. Η Τουρκία βαδίζει ταχύτατα προς εμφύλιο πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει λοιπόν να παρέμβει πάρα αυτά και χωρίς καθυστέρηση. Είναι αυτό επιταγή της ε, ανθρωπιάς. Ε, πρέπει να εμπλακούμε, φέρουμε ευθύνη και η τελευταία μου πρόταση κυρία Πρόεδρε, το κάτω-κάτω είναι και στο συμφέρον μας πρέπει να αποτρέψουμε την έξοδο γιατί αλλιώς θα υπάρξει νέα ε, μεταναστευτική ροή Κούρδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Εκ μέρους ε, των Σοσιαλδημοκρατών η κυρία Κάτι Πύρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ανατολική Τουρκία είναι πολύ ανησυχητική. Από τότε που ξαναξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΚΚ για τον τουρκικό στρατό, η κατάσταση επί τόπου έχει χειροτερέψει πολύ. Φανταστείτε να ζει κανεί στην Τσίζρα, στην Σινόπη, σε κάποια άλλη πόλη τη περιοχή. Ε, ε, στις αρχές Δεκεμβρίου εκεί ε, κηρύχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για πάρα πολλέ ώρε. Πάνω από 200.000 ε, άτομα χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια του. Ε, λαμβάνουν χώρα συγκρούσει και μάχε μέρα νύχτα ανάμεσα στον τουρκικό στρατό και του ε, αντάρτες που έχουν ε, στρατοπεδεύσει μέσα στι ε, πόλεις. Ε, όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τον πληθυσμό Να μην, μπορεί να, βγει, από το σπίτι σου για πάνω από 40 μέρε να σε παραστατικές οργανώσεις που τρομοκρατούν τον κόσμο, ένα μεγάλο αριθμό νεκρών στον άμαχο πληθυσμό, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Πώς είναι δυνατόν ένα 16χρονο παιδί να πεθάνει από αιμορραγία στο δρόμο χωρίς να μπορέσει ε, κανείς να τον ε, βοηθήσει. Ε, οι επιθέσεις του ΠΚΚ την περασμένη εβδομάδα ε, σκότωσαν αστυνομικούς και μέλη των οικογενειών τους. Δεν δικαιολογούνται. Γιατί όμως ε, να γίνονται επιθέσεις, ε, βίες επιθέσεις εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών. Πάνω από χίλια ακαδημαϊκοί στην Τουρκία ε, διώκονται επειδή υπέγραψαν μια, ένα κείμενο που ζητούσε ειρήνη. Πώς μπορούν αυτοί που, ζητούν την ειρήνη να κατηγορούνται για προδοσία. Ε, προφανώς κανείς δεν αμφισβητεί τον αγώνα της Τουρκίας εναντίον της τρομοκρατίας. Όμως αυτό που αμφισβητείται ε, είναι οι μαζικές ε, τιμωρίες ε, που δεν ε, κατευθύνονται εναντίον των συγκεκριμένων υπετίων αδικημάτων. Θα πρέπει να ζητήσουν να σταματήσει η σύγκρουση και να αρχίσει η ειρηνευτική διαδικασία. Θα πρέπει να αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορία και ε, θα πρέπει ο τοπικό πληθυσμό να στηριχθεί. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ για το ECR ο κύριος Μάρκ Ντεμεσμάκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, άκουσα τα οποία είπατε και συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες. Η πραγματικότητα είναι πως ε, ο τουρκικός στρατός ε, μετέτρεψε το Κουρδιστάν σε ένα λουτρό αίματος. Ολόκληρες ε, γειτονιές ισοπεδώνονται και λένε ότι έτσι σταματάνε την βία και εννοούν ότι γεμίζουν οι δρόμοι πτώματα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ο αυξανόμενος αυταρχισμός του Ερντογάν και του κόμματος του. Η προτεραιότητα δεν είναι να πολεμήσει το Ισλαμικό κράτος, αλλά να πολεμήσει τους Κούρδους και να αποκτήσει απόλυτη εξουσία και η δυτική σύμμαχη σιωπή. Καμία κριτική, καμία καταδίκη. Χρειαζόμαστε τον Ερντογάν για να σταματήσει τους πρόσφυγες. Και ντρέπομαι εγώ κύριε Χάν γι' αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το ανάστημα να υπερασπίσει τους Κούρδους. Έναν περήφανο λαό της ε, περιοχής, τον μοναδικό αξιόπιστο σύμμαχό μας κατά του Ισλαμικού κράτους, τον οποίο μαχαιρώνουμε στην πλάτη. Τι θα κάνει λοιπόν η Κομισιόν, επαναλαμβάνονται οι ενταξιακές ε, συνομιλίες, μα πρέπει να το κάνετε προϋπόθεση, κάντε προϋπόθεση την ειρήνευση δεν είναι σωστή η επιλογή που έχετε. Ευχαριστώ. Ο Αλεξάνδρ Γκραφ Λάμστοφ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία είναι τραγική. Την παρουσιάσατε με πλαστικά ε, χρώματα. Ε, σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς ε, να κατηγορήσει για πολλά την Τουρκία, την τουρκική κυβέρνηση, αλλά εκείνο που δεν μπορεί να την κατηγορήσει είναι ότι η ίδια ξεκίνησε αυτό αυτή την αντιπαράθεση. Το ΠΚΚ ήταν εκείνο το οποίο κατήγγειλε την κατάπαυση του πυρός ε, και την εκεχηρία δολοφονώντας δύο Τούρκους αστυνομικούς. Έτσι ξεκίνησε η όλη κατάσταση. Και αυτό που δεν εκτίμησε καλά το ΠΚΚ είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις στην Τουρκία ήταν ευγνώμονε για αυτή την εξέλιξη γιατί τους δόθηκε ευκαιρία να εξωθήσουν μια κατάσταση να επιδείξουν όλο και πιο αυταρχικό στυλ διακυβέρνησης. Αυτή η επίθεση έναντι των δύο πολιτικών έλαβε χώρα ανάμεσα σε δύο εκλογικούς γύρους στην Τουρκία ε, το κυβερνών κόμμα είχε χάσει την απόλυτη πλειοψηφία, την ανέκτησε, αυτό συνέβη και έκτοτε λοιπόν η κατάσταση έχει παγιωθεί. Ε, βεβαίως και πρέπει να ε, αναζωογονηθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Το ΠΚΚ οφείλει να αναγνωρίσει ότι ποτέ δεν μπορεί να νικήσει στρατιωτικά την Τουρκία σε συνεργασία με τη Συρία, με το Δημοκρατικό Κόμμα της ε, Συρίας, αν ενωθούν, ίσως ε, κάτι να καταφέρουν στην Ετεντολική Τουρκία, τουλάχιστον έτσι πιστεύουν. Αλλά εγώ σας λέω, αυτό δεν θα, το, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και έχει έρθει η στιγμή να το καταλάβει αυτό το ΠΚΚ. Αλλά και η κυβέρνηση στην Τουρκία. Και αυτή πρέπει να κατανοήσει ότι η αυτονομία είναι ένα πολιτιστικό αγαθό για τους Κούρδους είναι παραπάνω από αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν είναι μόνο οικονομικό το μέτρο. Είναι μια μορφή αυτοδιαχείρισης που θα πρέπει να τους εγκριθεί και όσον αφορά την ε, αυξανόμενη, την αυξανόμενη αυταρχική μορφή διακυβέρνησης. Η κυρία Πύρη τα είπε πάρα πολύ σωστά. Επόμενος ο κύριος Χατζηγεωργίου παρακαλώ, εκ μέρους της ΓΚΟΕ για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις έχω από τη Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία στην παρουσία του πρέσβη τη χώρα, όπου οφείλω να σα πω ότι ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν έριξε σχεδόν όλο το βάρο τη ευθύνη για το τι τρέχει στην νοτιοανατολική Τουρκία στο ΠΚΚ. Θεωρώ ότι αν μια περιοχή μισού εκατομμυρίου ανθρώπων βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό εδώ και δύο μήνες, αν αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στο ΠΚΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να το πιστέψουν. αν όμω συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε πρόκειται περί επανάσταση παρά περί τρομοκρατική ε, δραστηριότητας τόσων πολλών ανθρώπων. έχω λάβει προ λίγου μήνυμα από βουλευτή του ΧΑΤΕΠ, ο οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένος σε σπίτι στην περιοχή του σουρ βάλετε το σπίτι από τάγκ και από στρατιώτε και στέλνει το μήνυμα ότι ίσω είναι το τηλεφώνημα που έκανε, το τελευταίο τηλεφώνημα που κάνει στη ζωή του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που η Τουρκία οφείλει να αντιμετωπίσει και έχει μεγάλες υποχρεώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το μήνυμα να το δώσει καθαρά στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σκάκελερ για 1,5 λεπτό. Η κατάσταση στην Νοτιοανατολική Τουρκία είναι πολύ απογοητευτική. Είναι καταστροφική, άμαχοι σκοτώνονται κάθε μέρα σχεδόν. Ε, η κατάσταση όμως δεν είναι πολύ κακή μόνο στην, στην κουρδική περιοχή, αλλά σε όλη την Τουρκία. Ε, οι ακαδημαϊκοί έκαναν μια έκκληση ειρήνης. Είναι πραγματικά ήρωες. Και τι συμβαίνει, αντί να τους χειροκροτήσουν όλοι, τους απειλεί ο πρόεδρος Ερντοάν ακόμα και ένας αρχιμαφιόζος. Η ελευθερία τους απειλείται, η ελευθερία λόγου απειλείται και θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Εκεί όμως που οι πιο πολλοί συμφωνούμε νομίζω είναι ότι τα προβλήματα στην Νοτιοανατολική Τουρκία και στην Τουρκία συνολικά υπάρχουν, αλλά δεν συμφωνούμε όλοι ενδεχομένως για το τι πρέπει να κάνουμε Κατά την άποψή μου ήταν τεράστιο λάθος να ξεκινήσουν οι διαπραγμα... να μπλοκάρουν ένα-δύο κράτη-μέλη τις ε, διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας. Ε, γιατί αυτό ε, βοήθησε τον Ερντοάν στην εσωτερική του πολιτική και το χειρίστηκε με πολύ εφιός. Ας μην επαναλάβουμε αυτό το λάθος. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάντα ισχυρή σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιμένει. Το ίδιο και με την Τουρκία. Ασφαλώς θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία και για τους ε, πρόσφυγες. Όμως επουδενή δεν θα πρέπει να πουλήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν και ήδη πρόσφυγες. Ευχαριστώ για την ομάδα e Ο κύριος James Carver για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πώς μεταχειρίζονται οι Τούρκοι τους ε, Κούρδους ε, και στην Τουρκία αλλά και αυτούς που πολεμούν το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και Συρία είναι σκάνδαλο. Όλοι χαρήκαμε όταν σταμάτησαν οι εχθροπραξίες αλλά τώρα βλέπουμε πως ξαναρίχνουν λάδι στη φωτιά οι τουρκικές αρχές. Δεν φτάνει που επιτίθεται σε δημοσιογράφους και στην ελευθεροτυπία ο κ. Ερντογάν, αλλά τώρα επιτίθεται και στους Κούρδους. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμπεγνία μεταξύ των τουρκικών αρχών και του Ισλαμικού κράτους στην ε, περιοχή για να πολεμήσουν τους ε, Κούρδους. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των τουρκικών και των ευρωπαϊκών αρχών και περαιτέρω απόδειξη του ότι δεν πρέπει ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, ο κύριος Τεχράφ. Κύριε Πρόεδρε, οι δυτικέ αξίες, η ελευθερία, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν συμβάζονται με το Ισλάμ, με την Ισλαμιστική Τουρκία και το αποδεικνύει η Τουρκία κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα βάζουν τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή, μετά τους δημοσιογράφους και τώρα πολεμάνε τους ίδιους τους, τους το τέρας ε, της ε, Άγκυρας συνεχίζει τους ε, εκβιασμούς του. Ερωτώ τον κύριο Χάν, θεωρείτε πραγματικά πως τα εκατομμύρια πρόσφυγες που ήταν ασφαλείς στην Τουρκία ήρθανε με τον άνεμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σταματήσετε αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο συνέβη με τους Αρμένιους συμβαίνει τώρα και με τους ε, Κούρδους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο, δεν έχει καμία δουλειά η Τουρκία στην Ευρώπη, καταδικάστε τους και σταματήστε και τις διαπραγματεύσεις για ένταξη. Ένα μισή λεπτό. Τον λόγο έχει ο κύριος Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Ντεχράφ. Να πω κάτι σε εσάς είναι απαράδεκτο και αναξιοπρεπές να βάζετε στο ίδιο τσουβάλι εκατομμύρια μουσουλμάνους με τον ε, κύριο Ερντογάν ο οποίος παραβιάζει το δίκαιο και κάθε έννοια δικαίου δεν θα το δεχτούμε. Δεύτερον, είναι σωστό η τρομοκρατικές επιθέσεις ε, συναντούν αντίσταση και στην ε, Τουρκία και γεγονό είναι πως ο αντιπρόεδρος ο κύριος Τίμερμανς ε, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με την τουρκική κυβέρνηση για να μετριαστούν οι προσφυγικές ροές και γεγονός είναι πως περιέχει η συμφωνία αυτή περισσότερες διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Δυστυχώς επέλεξαν τα λάθος κεφάλαια έπρεπε να ξεκινήσουν από το 23 και το 24, το κράτος δικαίου και την ελευθερία, γιατί θα είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αποστολή της Κομισιόν να ξεκαθαρίσει πως ε, θα πρέπει να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία, το κάνουν αυτό, και πρέπει να πείτε ξεκάθαρα δύο λόγια στον Τούρκο Πρόεδρο για την πολιτική του γιατί εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι μέλη του ΠΚΚ. Είναι και θέμα δικής μας αξιοπιστίας να λύσουμε τα προβλήματα αυτά με τους ε, Τούρκους, αλλά δεν μπορεί να είμαστε τυφλοί και μουγκοί. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ. Η πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης ε, είναι όλο και πιο αυταρχική. 27 ακαδημαϊκοί διώκονται τελευταία Πολλοί δημοσιογράφοι επίσης. Εν τω μεταξύ, ο στρατός ε, πολεμάει το ΠΚΚ, το οποίο είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ταυτόχρονα εκατοντάδες άμαχοι χάνουν τη ζωή τους, υπάρχει ε, απαγόρευση κυκλοφορίας και περιορισμός των πολιτικών ελευθεριών. Οι τουρκικές ε, αρχές ε, εξακολουθούν να θεωρούν τους Κούρδους ως τη μεγαλύτερη απειλή και όχι τον Άισις. Η Τουρκία ε, προσπαθεί να αποφύγει τη δημιουργία κουρδικού κράτους αντί να προσπαθεί να πολεμήσει τον, το Ισλαμικό κράτος. Ταυτόχρονα ε, δεν συνεργάζεται επαρκώς για να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη. Θα πρέπει η αρχή οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων να ζητήσουν από την Τουρκία να εφαρμόσει τις ε, υποσχέσεις της και να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τον Ερντοάν. Oh, Κύριε Λάμπστορφ, ο κύριος Λάμστορφ έχει μπλε κάρτα για τον κύριο Τάνοκ. Δέχεστε. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά, λέει ο κύριος Λάμπστορφ, Λοιπόν, ε, άκουσα πολύ προσεκτικά. Ε, υπάρχει υποτροπιασμός ε, στον αυταρχισμό, σύγκρουση της τουρκικής κυβέρνηση με σουνίτες παραστρατιωτικούς υπάρχει η επαναπροώθηση προς τη Συρία, υπάρχει θεοκρατικό αυταρχικό στυλ διακυβέρνησης της τουρκικής κυβέρνησης. Charles, σε ρωτάω, η συντηρητική της Μεγάλης Βρετανίας ήταν πάντα διαπρίσει κήρυκες ε, της ε, σωστής διακυβέρνησης Τουρκία και υποστηρικτές του Ερντογάν. Άλλαξε κάτι. Και εγώ στην προηγουμένη συζήτηση ε, σε είχα ρωτήσει αν είσαι υπέρ του να ανασταλεί οικονομική βοήθεια στην Τουρκία και μου είχε δώσει μια απλή απάντηση. Θα σου δώσω και εγώ την απλή απάντηση ότι η επίσημη θέση μας είναι ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, αυτή τη στιγμή υφίστανται σημαντικές ανησυχίες για την αλλαγή πορείας που έχει δείξει ε, η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι πολύ μακριά από το να είναι ικανή να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Βρετανία θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Σχάγε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ η συμφωνία για την μετανάστευση που έσπευσε να υπογράψει ο κύριος Τίμερμανς φαίνεται να είναι ο λόγος για τον οποίο η επικίνδυνη κατάσταση ε, αντιμετωπίζεται με εκοφαντική σιωπή από τα κράτη-μέλη της Ένωσης και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δούμε πάρα πολλά ζητήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση του ΑΚΠ να επανέλθει στην ενετική διαδικασία με το ΠΚΚ και να σταματήσουν οι δυσανάλογες ε, παράπλευρες απώλειες αμάχων. Ποτέ δεν δικαιολογείται η τρομοκρατία και η δημοκρατική πορεία των Κούρδων είναι η βασική εναλλακτική που πρέπει να προκύψει. Και όταν οι πανεπιστημιακοί ζητούν ε, να σταματήσει η βία είναι ελευθερία τους. Πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε έναν αξιόπιστο εταίρο στην Τουρκία που είναι χώρα του ΝΑΤΟ και να γίνει ενεργό μέλο του συνασπισμού κατά του Ισλαμικού κράτους. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα των στόχων μας. Και να είμαστε προσεκτικοί ή να μην χρησιμοποιηθεί η αντιδρομοκρατία ως δικαιολογία για να περιοριστούν τα δικαιώματα και ελευθερίε των ανθρώπων στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βερζιά. Για ένα λεπτό. Εδώ και πάνω από ένα μήνα ο τουρκικός ε, στρατός ε, επιχειρεί με βία στην Ανατολική Τουρκία, στην μια περιοχή που έχει πλειοψηφία κουρδικού πληθυσμού. Ε, το ΧΑΝΤΕΠΕ καταπιέζεται, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και πανεπιστημιακοί ακαδημαϊκοί που, για παράδειγμα, υπέγραψαν μια έκκληση ειρήνης δεν είναι αιτία του ΠΚΚ, η ε, δεν είναι το ΠΚΚ αιτία της σύγκρουσης όπως λέει η Άγκυρα. Ε, πολλά παιδιά, πολλές ε, οικογένειες ε, ε, φίστανται τα αποτελέσματα. Μέχρι και πεντάχρονα παιδιά έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατίες. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί έστω και μονομερό, έτσι ώστε τα μέρη να γυρίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να υποχρεωθεί η τουρκική κυβέρνηση να ξαναξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων, είτε είναι πολιτικά είτε είναι θρησκευτικά, θα πρέπει να αναγνωριστούν. Θα πρέπει να, σταματήσει ή, να σταματήσουν οι διακρίσει. Πιστεύω ότι είναι πήγον να διοργανώσουμε ε, μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Τουρκία και να την αποστείλουμε εκεί. Ευχαριστώ. Valero, Κυρία Βαλέρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, τα κτίρια πέφτουν, οι εκκλησίες καταστρέφονται βομβαρδίζονται. Αυτό, αυτό δήλωσε ο, ο, ο κύριος Ερντοάν, ο πρόεδρος Ερντοάν είπε ότι θα καταστρέψουν ακόμα και οποιαδήποτε κτίρια ή εκκλησίες ε, στις οποίες κρύβονται μαχητές του ΠΚΚ. Ταυτόχρονα θα χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άμαχοι. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Γιατί χάνουν κάθε μέρα. Μεταξύ αυτών πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά. Μας έχουν στείλει βίντεο που δείχνουν τι συμβαίνει στην περιοχή. Οι πληροφορίες μας ε, αποδεικνύουν ότι η κατάσταση είναι διαφορετική από αυτήν που καταγγέλει ο Ερντοάν. Χρειάζονται τόσοι στρατιώτες για να ε, καταστήλουν μια γριά γυναίκα. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ο Ερντοάν δεν τηρεί τις υποσχέσεις του να σταματήσει τις ροές των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ο κ. Φερόν για ένα λεπτό. Θα σας πω ένα μυστικό. Πριν από μερικά λεπτά ε, ήμουνα στην συνάντηση της, ε, Επιτροπής με την Τουρκία. Εδώ και δέκα μήνες δεν είχαμε ε, συναντηθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε γιατί. Γιατί κάθε φορά που ήταν να συναντηθούμε, ε, είναι, κάθε φορά που συναντιόμαστε είναι παρόν ο, ο, ο πρέσβης της, Ευρωπαϊκής, της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος ε, μιλάει πολύ περισσότερο οποιοδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σαν να είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως όχι ως μέλος αλλά μέλος, μέσω των πράξεών της. Ε, κάθε μέρα στην Τουρκία λαμβάνει η χώρα ε, μια επίθεση ή κάποιο πεθαίνει, κάποιο χάνει τη ζωή του. Είναι συνεχώ στην επικαιρότητα. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τον κουρδικό λαό με την Τουρκία. Ε, υπό την κάλυψη του αγώνα εναντίον του Ισλαμικού κράτου, η Τουρκία αποφάσισε να πολεμήσει εναντίον τη αντιπολίτευσή τη. Αυτό για μία ακόμα φορά αποτελεί ε, απόδειξη ότι δεν είναι μια ακομα φορα αποτελει αποδειξη οτι δημοκρατία που έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστώ για μισή λεπτό ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα επαναλάβω. Εγώ είμαι μεταξύ των φίλων και υποστηρικτών της Τουρκίας και της ενίσχυσης της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία είναι πρώτα απ' όλα κατά των τουρκικών συμφερόντων. Η βία, η κλιμάκωση της βίας στην νοτιοανατολική Τουρκία είναι ένας πραγματικός κίνδυνος που πρέπει να σταματήσει. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε πολιτικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των Κούρδων για να επανέλθουν στο σημείο στο οποίο είχαν ε, φτάσει με σημαντικές πρόοδους στην ειρηνευτική διαδικασία. Όλα αυτά χάθηκαν τώρα και φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο θα είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση. Θα επαναλάβω πως πρώτα απ' όλα το συμφέρον της Τουρκίας είναι να αποτρέψει την περαιτέρω αποσταθεροποίηση και κλιμάκωση της βίας που μπορεί να καταλήξει σε εμφύλιο πόλεμο. Και πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο να καταδεκάσουν χωρίς εξαίρεση όλα τα λάθη των εταίρων μας και της Τουρκίας. Γιατί είναι μακροπρόθεσμοι οι εταίροι μας, πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους και έχουμε κοινέ προκλήσεις και αξίες, αλλά πρέπει να έχουμε αυτές κοινέ αξίες και στο μέλλον και να έχουμε το θάρρος ε, να ζητήσουμε από την Τουρκία άμεση κατάπαυση του πυρός, ειρηνευτική διαδικασία και άμεσες επισκέψεις στο σημείο εκείνο στο οποίο δεν επιτρέπεται να πάει κανείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να παραμένετε εντός του χρόνου. Πριν δώσω λόγο στον κύριο Μαριά, να πω πως υπήρξε μια μπλε κάρτα από έναν συνάδελφο που έχει ήδη μιλήσει και ξέρω πως πολλοί συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν στο τέλος της συζήτησης στο KTI, οπότε αν συμφωνείτε θα περάσω στον επόμενο μιλητή. Λοιπόν, ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να πάψει να εθελοτυφλεί μπροστά στις κατάδυλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του κουρδικού λαού, στις οποίες προβαίνει ο τουρκικός στρατός στις νότιο-ανατολικές επαρχίες. Οι βιαιότητες του τουρκικού στρατού έχουν οδηγήσει 200.000 ανθρώπους, κατά πλειοψηφία Κούρδους, να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους ολόκληρες πόλεις έχουν αποκλειστεί και οι κάτοικοι καθυλώνονται σε κατάσταση απαγόρευσης κυκλοφορίας. εκλεγμένοι δήμαρχοι και πολιτικοί του φιλοκουρδικού κόμματος χαντεπέ διώκονται ποινικά ενώ άλλοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή σε ένα όργιο αυταρχισμού από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης. σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης η κυβέρνηση της τουρκίας θέλει να έχει ολοκληρώσει αυτή τη δίθεν αντιτρομοκρατική επιχείρηση μέχρι την άνοιξη προειδοποιούμε ότι η ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτοφανούς έξαρσης στρατιωτικής βίας και ο χρόνος που δίνεται να επέμβει στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου είναι περιορισμένος. ζητούμε λοιπόν από την ευρωπαϊκή ένωση να λάβει άμεσα μέτρα κατά της τουρκίας και να της κλείσει την πόρτα προς την ευρώπη αντί να θοπεύει την άγκυρα και να ανέχεται τα ανατολίτικα τερτύπια της. ευχαριστώ. Uh, Κοιτάξτε, ένας συνάδελφος έχει ζητήσει μπλε κάρτα, αλλά είστε και στο KTI. Δεν είστε στο KTI. Ήσασταν στον κατάλογο μου. Εντάξει, να σας δώσω τότε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα, εάν το δέχεται ο κύριος Μαριάς. Ωραία. Κύριε συνάδελφε, αντιλαμβάνομαι ότι είστε Έλληνας και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει με κάποιον τρόπο και να απευθύνει μια επιστολή προς τον πρόεδρο Ερντογάν για να μεσολαβήσουμε στις συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης Τουρκίας και των ακροσώπων των Κούρδων. Γιατί ξέρετε η σταθερότητα της Τουρκίας, αποσταθεροποίηση της Τουρκίας θα σημαίνει αποσταθεροποίηση της Ελλάδας και της Ευρώπης. Κύριε συνάδελφε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρει τρόπους προκειμένου να αναγκάσει την Τουρκία επιτέλους να εφαρμόσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό πρέπει να γίνει με τη λήψη μέτρων διότι μέχρι στιγμή αυτό που γίνεται είναι να θοπεύει η ευρωπαϊκή ένωση την τουρκία να ανέχεται τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο κατά των κούρδων αλλά και κατά των άλλων υπολείπων τούρκων πολιτών την ανέχεται που έχει παραβιάσει το διεθνέ δίκαιο και κατέχει αυτή τη στιγμή το 37% τη Κύπρου. Την ανέχεται που έχει στρατεύματα μέσα σε μια χώρα που είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ληφθούν μέτρα για να καταλάβει η τουρκία τι πρέπει να κάνει. ευχαριστώ. It 30 seconds δευτερόλεπτα έχετε παρακαλώ για τις απαντήσεις σας. Σεβαστείτε το. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Για ένα λεπτό ο κύριος Χουαρίστια Μπάντς. Ε, δεν μου αρέσει όταν χρησιμοποιούμε την κατάσταση των προσφύγων ε, που κατά εκατομμύρια αποδρούν από τις ε, συγκρούσεις ε, σε αυτές εκείνες τις περιοχές. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία ε, είναι τα αίτια. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δολοφονεί κατά Τούρκους, Κούρδους και η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τα αυτιά της. Αυτό είναι απόλυτο απαράδεκτο. Κύριε Επιτροπέ, πέραν των λόγων και των προθέσεων, οι πράξεις των κρατών μελών, ε, οι σχέσεις με την Τουρκία, ε, η εγκατάλειψη των Κούρδων είναι προφανής. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε σιωπηλοί ενώπιον της ε, μαζικής και συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του τουρκικού κράτους. Ευχαριστώ. Κύριε Λάμπερτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πρώτη φορά πήγα σε αυτήν την περιοχή της Τουρκίας πριν από 15 χρόνια. Είχε στρατιωτικό νόμο, είδαμε εγκαταλειμμένα χωριά, καταπίεση και τώρα ξανά εκεί επιστρέψαμε. Και όπως είπαν και άλλοι χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία ειρηνευτικής διαδικασίας. Και από την κυβέρνηση που δεν μπορούσε να δεχτεί ένα ειρηνικό κουρδικό κόμμα το οποίο ξεπέρασε το εκλογικό όριο του 10% στις τελευταίες εκλογές. Αλλά είδαμε και συμμάχους του ΝΑΤΟ να επιτρέπουν τις ε, τουρκικές επιθέσεις κατά του ΠΚΚ σε αντάλλαγμα για πρόσβαση σε τουρκικές βάσεις για να επιτεθούν στο Ισλαμικό κράτος. Το ΠΚΚ δεν είναι το Ισλαμικό κράτος. Ναι, έχει επιτεθεί σε αμάχους και πρέπει να το καταδικάσουμε. Αλλά πρέπει αυτή την σημαντική ε, δυσαρμονία να την δουν οι κυβερνήσεις για να επανέλθουμε στην ειρηνευτική διαδικασία και να επικεντρωθούμε στην πραγματική απειλή. Ευχαριστώ. Βάιντεν Χόλτσερ για ένα λεπτό. Η Τουρκία είναι μια υποψήφια χώρα και ξαναξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να θέσουμε και κρίσιμες ερωτήσεις για τα θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων είναι πολύ ανησυχητικές και αφορούν το κουρδικό. Η τωρινή κυβέρνηση θεωρεί ότι θα λύσει το πρόβλημα με την βία και ότι έχει μια εξουσιοδότηση εν λευκό. Μετά από μια φάση συνομιλιών έχουμε ξανά εχθροπραξίες. Δεν είναι προς το συμφέρον μας αυτό. Κύριε Επίτροπε, σας ζητώ να υπενθυμίσετε στους Τούρκους πως δεν είναι προς ε, το συμφέρον μας αυτό και το δικό του συμφέρον. Θα πρέπει η Ευρώπη να απευθύνει έκκληση και στις δύο πλευρές να αναστείλουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διαμεσολαβητής. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να ακολουθεί το παράδειγμα της Βορείου Ιρλανδίας όπου όλοι οι αντιμαχόμενοι κατέληξαν στην τραπέζα διαπραγματεύσεων ακόμα και αυτοί που τότε τους έλεγαν τρομοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριος Χρυσόγονος για ένα λεπτό το καθεστώς ερντογάν καταδικάζει στην πείνα τους πολίτες στην νοτιοανατολική τουρκία μέσω των απαγορεύσεων κυκλοφορίας που έχει επιβάλει επί εβδομάδες ολόκληρες. επιτίθεται εναντίον κουρδικών πόλεων και χωριών με βαριά όπλα και καταπατάει συστηματικά τα δικαιώματα των κατοίκων τους στη ζωή την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια καθώς και την απαγόρευση των βασανιστήριων. η προμελετημένη αυτή σφαγή και η εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων κούρδων από τις αιστείες τους παραβιάζει τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και το τουρκικό σύνταγμα. το καθεστώς ερντογάν αρνείται την πρόσβαση ανεξάρτητων παρατηρητών στις κουρδικές περιοχές και καταδιώκει πολυάριθμους διανοούμενους που έχουν καταγγείλει τις απάνθρωπες πρακτικές του. με την ανοχή της απέναντι στα εγκλήματα αυτά η ευρωπαϊκή ένωση προδίδει τις ιδρυτικές της αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. η προσπάθεια κατευνασμού του καθεστώτος ερντογάν είναι λάθος. η μόνη γλώσσα την οποία μπορεί να καταλάβει είναι η γλώσσα των πολιτικών και οικονομικών κυρώσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλοί άξιοι συνάδελφοι περιέγραψαν πιστά την κατάσταση που υπάρχει στην νοτιοανατολική Τουρκία μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων δεν θα επαναλάβω τα λόγια τους. Θα επαναλάβω όμως τα λόγια του Σουλεϊμάν Ντεμιρτάς, του Προέδρου του ΧΑΝΤΕΠΕ. Το ΧΑΝΤΕΠΕ είναι το κόμμα που υποστηρίζεται μαζικά από την κουρδική μειονότητα και όχι μόνο από αυτήν. Το, το ΧΑΝΤΕΠΕ δεν προκάλεσε τον πόλεμο. Το ΧΑΝΤΕΠΕ δεν καθοδηγεί τη σύγκρουση, δεν την ελέγχει. Από μία πλευρά βρίσκεται το χέρι του Προέδρου Ερντογκάν, από την άλλη βρίσκεται το χέρι του ΠΚΚ. Αυτά είπε ο Πρόεδρος Ντεμιρτάς θα πρότεινα στο σώμα και στον επίτροπο ΧΑΝ να καλέσουμε την τουρκική εθνοσυνέλευση να κάνει μια γενναία πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στην κατάπαυση του πυρό και στην ειρηνευτική διαδικασία. Και θέλω να προσθέσω ότι αν χρειάζεται θάρρο για να πάρει τα όπλα να προστατευτεί απέναντι στην ασύμετρη κυβερνητική βία, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερο θάρρο να ξεπεράσει τι προκλήσει και να οδηγήσει στην ειρηνευτική διαδικασία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, εγώ επιβεβαιώνω ότι υπάρχει αυτή η έκκληση από πλευρά διανομένων Ιταλών ε, και επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει μία προμελετημένη σφαγή. Σε πολλές πόλεις ε, η απαγόρευτη κυκλοφορία σχεδόν και μήνες, δεν υπάρχουν τρόφιμα. Επίσης ε, έχουν βομβαρδιστεί ακόμα και πόλεις όπου δεν ήταν καν πολιορκημένες. Αυτοί που υπογράφουν αυτή την έκκληση θεωρούνται συνομότες και συνεργοί των τρομοκρατών. Υποτίθεται έχουν παραβιάσει το τουρκικό σύνταγμα. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι απλά μία πρόφαση. Ο στόχος είναι να σφαγιαστεί ένας λαός ο οποίος όμως είναι τμήμα αυτής της χώρας. Χιλιάδες Τούρκων προσβλέπουν στη διαμεσολάβηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση που διέκοψε ο Ερντογάν. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ε, απαντώντας σε μια δική μου ερώτηση, η κυρία Μογκερίνη μου είπε ότι ο Ερντογάν είναι σύμμαχός μας για τα θέματα των προσφύγων και κατά του ISIS. Αυτή η επιχειρηματολογία δεν στέκεται μα ούτε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάνι, θα έχει μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε κύριε Σπινέλη. Ωραία, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πράγματι, έχετε εμπλακεί προσωπικά σε αυτό το θέμα και το εκτιμώ. Δεν πιστεύετε ότι θα ήταν σημαντικό να διατηρήσουμε θεσμικές επαφές. Για παράδειγμα, η κοινοβουλευτική συνέλευση του ε, ε, ΝΑΤΟ θα μπορούσε Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε έρθει σε επαφή όχι μόνο με την ύπατη εκπρόσωπο αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη και πάνω απ' όλα με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Λόπες. Η κλιμάκωση της ε, βίας στην Τουρκία συνεχίζεται. Πρόκειται για μια βία που επιδεινώνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Ε, έχει μάλιστα ένα χαρακτήρα συλλογικής τιμωρίας του κορδικού πληθυσμού με δεκάδες ε, χιλιάδες μετακινούν πληθυσμού, εκατοντάδες νεκρούς άμαχους, εκατοντάδες άτομα τα οποία συλλαμβάνονται και κρατούνται χωρίς λόγο. Ε, θα πρέπει να ζητήσουμε ανακοχή, ε, θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ε, που σταμάτησαν ξαφνικά το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα να υπενθυμίσουμε μια στιγμή που εντείνουμε τη συνεργασία μας με την ε, Τουρκία, να υπενθυμίσουμε, λέω, στην Τουρκία ότι αυτή η συνεργασία δεν μπορεί επουδενή να αποτελέσει αντάλλαγμα για οτιδήποτε άλλο, ιδιαίτερα ε, για την ε, ενόψη της κρίσης με, το, με τους πρόσφυγες. Εν πάση περιπτώσει η κατάσταση σήμερα στην Νοτιοανατολική Τουρκία είναι απαράδεκτη και αυτό θα πρέπει να δηλωθεί πανηγυρικά. Υπάρχει αίτημα για μπλε κάρτα κύριε Λόπεθ. Τη δέχεστε. Ο κύριος Μπονάνο. Τη δέχεστε. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το συνάδελφό μου το εξής. Πιστεύει και εκείνος ότι η Τουρκία σίγουρα δεν συμπεριφέρεται σωστά, αλλά δεν συμπεριφέρεται σωστά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, μερικοί λένε δεν συμπεριφέρεται σωστά αιώνε η Τουρκία, αν δει κανεί την ιστορία τη. Είναι λοιπόν σωστό το ότι η Ευρώπη τη έδωσε 10 δι και λέει θα της δώσει άλλα 3 δι. Ε, όταν κάποιο δηλαδή συμπεριφέρεται χάλια, του δίνουμε και λεφτά από πάνω. Ε, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά της ε, Τουρκίας ε, πολλές φορές, αλλά όταν δίνουμε χρήματα δεν τα δίνουμε στην κυβέρνηση και στο κράτος, ε, τα δίνουμε αυτά τα χρήματα για τους πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή ζουν και υποφέρουν στην Τουρκία. Πρόκειται για σύρους πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά δε, την συμπεριφορά, ούτε, με, ούτε και η δική σας συμπεριφορά πολλές φορές δεν μ' αρέσει, αλλά σέβομαι αυτά που λέτε και αυτά που κάνετε. Um, Να δώσω τώρα τον λόγο σε κάποιους ομιλητές αλλά πριν από το KTI περνάμε στον κύριο Μπενιφέ για ένα λεπτό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου στους ε, σοσιαλιστές ταντέλφους οι οποίοι προηγήθηκαν στο να καταγγείλουν αυτή την ε, τραγική κατάσταση που διαδραματίζεται εδώ και αρκετό ε, νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Αυτά που διαδραματίζονται δεν μπορούν να παραμείνουν απαρατήρητα από πλευράς Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η βία υπάρχει κίνδυνος να μετεξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο. Κατόπιν τούτου, η διεθνή κοινότητα οφείλει να στρέψει την προσοχή τη προ αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πολλού ε, εκτοπιστέντε, 300.000 περίπου. Ε, Ω εκ τούτου, ε, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από την κυρία Μογγερνή στην επόμενη επίσκεψή της στην Άγκυρα. Όσον αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία, πρέπει να υπάρξει το των δυνατόν κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική διαδικασία. Εμείς έχουμε στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία για τους Κούρδους και τώρα δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από διάφορα που είναι η προσφυγική κρίση ε, για να κλείνουμε τα μάτια σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη διαδικασία Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο σε εννέα ομιλητές από όλες τις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε όλοι ε, στην παρέμβασή σας σε ένα λεπτό. Σρόιβοντα παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως η Τουρκία αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα σεβαστεί την Ένωση και ότι δεν θα εκμεταλλευτεί την περίσταση για να προωθήσει τα πολιτικά της συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή ε, όμως ε, οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων ε, έχουν τραγικές συνέπειες. Οι απαντήσεις του πρέσβη ε, δείχνουν όμως ότι ο τουρκικός ε, στρατός ε, ε, συγγνώμη, ισχυρίζεται ο πρέσβη τη Τουρκία ότι ο τουρκικό στρατό δράει νομίμω, αλλά εμεί δεν πρέπει να μείνουμε σιωπηλοί. Ποιο Καπούτο, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, από το Δεκέμβριο του 2015 διάφορες περιοχές της νοτιοανατολικής ε, Τουρκίας ε, πλήττονται ε, τουλάχιστον τέσσερις φορές την ημέρα. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι πλέον σε θέση να αγοράσουν τρόφιμα ούτε φάρμακα. Είμαστε λοιπόν ανήσυχοι και για τις συλλήψεις των ακαδημαϊκών που έγραψαν μια έκκληση για την ειρήνη. Στην νοτιοανατολική Τουρκία υπάρχουν παραστρατιωτικές ομάδες και αυτοί απειλούν τους υπογράφοντες στην έκκληση. Για πρώτη φορά έχουν δολοφονηθεί πάρα πολύ άμαχοι. Ε, το όλο θέμα είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε μια χώρα η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνω με τα λόγια του Κάνουν Ντάρ ενός ε, διευθυντή εφημερίδας ε, της αντιπολίτευσης που απευθύνεται στον κύριο Ρέντσι και του λέω ότι δεν πρέπει κανείς να αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία απλώς και μόνο ως αντάλλαγμα για τις προσφυγικές ροές. Αυτά είχα να πω. Ο κύριος Ζαμπάσκι. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην Ουτο-Ανατολική Τουρκία υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Εξάγεται εδώ και δεκαετίες και τώρα ξαναφούντωσε. Η κυβέρνηση αυτή καταλαμβάνει παρανόμως ε, εδάφη της Συρίας ε, και του Ιράκ και την Κύπρο εδώ και δεκαετίες. Προβαίνει σε εθνικές ακαθαρίσεις και γενοκτονία στις ε, κουρδικές περιοχές και στο Ιράκ και στη Συρία. Αυτές είναι οι σωστές λέξεις και εκπλήσωμε που υπάρχουν συνάδελφοι εδώ μέσα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση διέπραξε αυτοκτονία μετά τις εκατομμύρια που υποσχέθηκε γιατί περί αυτοκτονίας πρόκειται και αυτά τα οποία κάνει η τουρκική κυβέρνηση είναι γενοκτονία. Πρέπει να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία δεν έχει καμία δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό κυρία Σακόραφα. Κύριοι συνάδελφοι, η Τουρκία, η Τουρκία φλερτάρει με τον αυταρχισμό. Ο Ερντογάν με την ανοχή της Ευρώπης χτίζει την σύγχρονη τουρκική αυτοκρατορία του πάνω σε πτώματα Κούρδων αμάχων και στη δυστυχία εκατομμυρίων προσφύγων, πάνω στα συντρίμμια της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, πάνω στην ανυπαρξία ελευθερίας έκφρασης, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ελευθερία του τύπου και με μαζικές εκαθαρίσει στη δημόσια διοίκηση, συλλήψεις και κατηγορίες για εθνική προδοσία αντιφρονούντων, ακαδημαϊκών και Κούρδων πολιτών και πολιτικών. Οι απαγορεύσει κυκλοφορία, η στρατιωτική και αστυνομική βία δημιουργούν πόλει φαντάσματα με εκατοντάδε χιλιάδε εκτοπισμένου η τουρκία αδιαφορεί και για το σχέδιο δράσης που συμφωνήσατε στο προσφυγικό και για τους διακινητές. 31.000 πρόσφυγες, κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν το Αιγαίο αυτό το μήνα με 8 και 9 μποφόρ. Ποιος λοιπόν σε αυτή την αίθουσα μπορεί να υποστηρίξει ότι η κατάσταση αυτή παραπέμπει σε ασφαλή χώρα. Από αυτό το βήμα, κύριοι συνάδελφοι, καλώ την ύπατη εκπρόσωπο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίε ώστε να επιστρέψουν οι δύο πλευρέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να σταματήσει αυτό το σπιράλ βία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, γνωρίζουμε ότι, όλα σας συμβαίνουν ε, εκεί ε, δεν είναι απλώς μια μάχη εναντίον της τρομοκρατίας. Έχουμε συλλήψεις ε, διανοουμένων, κατοντάδες αμάχους νεκρούς, ε, διώξεις δημάρχων κλπ. Ε, μας το εξήγησαν οι δήμαρχοι του, του, της Μάντριν, του Διαρμπακύρ κλπ. Υπάρχουν εξηγήσει μας ε, για την στάση αυτή και οι μαρτυρίες των μη κυβερνητικών ανανόσεων τα επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε τα μάτια μόνο και μόνο για να το θέμα των προσφύγων. Ζητώ κύριε Επίτροπε, απαιτώ για την ακρίβεια, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμουν αμέσως. Ε, δεν αρκούν μόνο τεχνικές συναντήσεις ε, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει ήδη να σταλεί ένας ειδικός εκπρόσωπος στην Τουρκία για να πραγματικά να κηρυχθεί πραγματική ανακοχή. Τώρα για ένα λεπτό και παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Κύριο Καστάλτο. Πόσο κοστίζει και με τι νόμισμα πληρώνει κανείς ε, για να αποφευθεί η σύγκρουση με την Τουρκία για την προσφυγική κρίση. Πληρώνει κανείς με ευρώ, με αίμα και με αναξιοπρέπεια. Τα ευρώ τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, ελπίζοντας ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Το αίμα σε μεγάλο, μεγάλες ποσότητες το καταβάλουν οι Κούρδοι που είναι πολίτες ε, ενός κράτους, ε, όμως δεν αντιμετωπίζονται ως πολίτες την ε, έλλειψη αξιοπρέπειας. Αυτή την παρουσιάζουν οι ε, δικές μας, τα δικά μας τα όργανα, γιατί δείχνουν ανοχή απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία ποδοπατά όλες τις ελευθερίες. Και αυτό ισχύει για τη μειονότητα των Κούρδων. Τώρα λοιπόν συλλαμβάνουν ακόμα και δημοσιογράφους και καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτά όλα δεν είναι σωστά μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Πώς ακόμα θα ανεχθούμε. Δυστυχώς ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή και λέει θα δώσω τώρα για ένα λεπτό το λόγο στον κύριο Συναδινό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κατάσταση στην νοτιοανατολική τουρκία καλύπτεται από ένα πέπλο μυστικότητα και σιωπής δυστυχώ, και αυτό οφείλεται στην ανοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. τα δυτικά μέσα ενημέρωση αναπαραγάγουν μόνο ειδήσει που αφορούν σε απώλειε των τουρκικών δυνάμεων ασφαλεία, αποκρύπτοντας επιμελώς τι αναφορές στα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητας που διαπράττει το καθεστώς του αιμοσταγού ερντογάν. η γεωγραφική θέση των μαχόμενων για το δικαίωμα στη ζωή και ευημερία κούρδων αποτελεί δίωδο και γέφυρα για τι παράνομε πράξει και δοσοληψίε μεταξύ τη τουρκία και των τζιχαντιστών του ισλαμικού κράτου. η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να σχεδιάσει πολύ προσεκτικά τι γεωστρατηγικέ και γεωπολιτικέ τη κινήσει σε μια σκακέρα όπου υπάρχει τεράστια σύγκρουση συμφερόντων μα κυρίω ογκοδέστατη συγκέντρωση αντιμαχόμενων παρατάξεων. το χάο που επικρατεί μεταξύ των κούρδων τη τουρκία συρίας και ιράκ του ντάεσ των ουαχαμπιτικών ομάδων σιητών σουνιτών χριστιανών και τη φανερή ή μυστική ανάμειξη των ξένων δυνάμεων θα οδηγήσει μοιραία σε μια σύραξη με παγκόσμιες διαστάσεις. ευχαριστώ. Η... η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να χαρακτηρίσει όλο το κουρδικό κίνημα ως τρομοκρατικό ε, θέλει να πείσει την κοινή γνώμη ότι αυτό ισχύει. Όμως ε, για τους Κούρδους ε, η, η ειρήνευση απομακρύνεται κάθε μέρα που περνάει. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Κούρδους και την τουρκική κυβέρνηση έχουν σταματήσει. Παρόλο ότι στην αντιπολίτευση υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν την ενευτική διαδικασία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει την Τουρκία να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Παρόλο ότι πολλοί πιστεύουν πως ε, το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε για να μας βοηθήσει η Τουρκία στο προσφυγικό είναι να τους επιτρέψουμε να λύσουν το κουρδικό όπως επιθυμούν. Όμως μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία διαπραγματεύεται την ένταξή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλήσουμε στα ε, ανθρωπιστικά ε, προβλήματα. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής, το Κετσιάκη, και ζητώ συγγνώμη από όσους δεν μίλησαν, ο κύριος Παπαδάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια στις πραγματικότητες και να γίνουμε πιο ειλικρινείς μεταξύ μας σε σχέση με την Τουρκία. Δεν σημαίνει επειδή γίνονται εκλογές στην Τουρκία ότι είναι και δημοκρατική χώρα. Συνεχίζει να κατέχει το 38% της Κύπρου, διώκει τους αντιφρονούντες, φυλακίζει, συνεργάζεται με το ISIS και στέλνει πρόσφυγες στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Και τώρα που μιλάμε πραγματοποιεί γενοκτονία σε βάρος του κουρδικού λαού και όχι σε βάρος του ΠΚΚ αυτήν η τουρκία θέλετε για εταίρο λόγω του προσφυγικού να κλείνετε τα μάτια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ένας είναι ο δρόμος. Πραγματική εκδημοκρατικοποίηση της Τουρκίας. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει ακολουθώντας τον κατάλληλο δικό χάρτη από την Ευρώπη, χωρίς εκτόσεις για εξυπηρέτηση οποιοδήποτε άλλο συμφερόντο. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Επίτροπος για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την συζήτηση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για να σχηματιστεί, να εδρεωθεί μια γνώμη. Μου υπενθυμίσατε πως ε, την Δευτέρα ο κ. Στυλιανίδης και εγώ θα πάμε την Δευτέρα για, στην Άγκυρα για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και οπωσδήποτε θα θίξουμε το θέμα αυτό. Και οπωσδήποτε οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όσον αφορά τα κεφάλαια 23 και 24, αλλά είμαστε σε μια φάση της ε, προετοιμασίας και οποιοδήποτε ασχολείται λίγο με αυτά τα πράγματα γνωρίζει ξεκάθαρα πως την προετοιμασία αλλά και στην διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων το μεγαλύτερο ε, εργαλείο που έχουμε στην ε, διάθεσή μας είναι ακριβώς να ασκήσουμε κάποια επιρροή και είναι ακριβώς και η Λιδία Λίθος για να δούμε πόσο σοβαρά τα παίρνει αυτά τα πράγματα η τουρκική κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς εξετάζουμε και βεβαίω η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατή όταν κάποιο συμφωνεί με τις αρχές μας, τις πεπιθήσει μας και ε, το νομικό μας οικοδόμημα. για ε, διαπραγματεύσει δεν είναι για να προσεγγίσουμε τις ε, θέσεις μας, είναι για να προσεγγίσει η Τουρκία τις ευρωπαϊκές αξίες και να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ακριβώς αυτό είναι ο ισχυρότερος μοχλός που έχουμε στην διάθεσή μας και θεωρώ πως ε, εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ε, Κούρδους ε, στην Τουρκία γι' αυτό χαίρομαι για το ότι υπάρχουν και κάποιοι Τούρκοι δήμαρχοι εδώ πέρα οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν μαζί μας και να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες από πρώτο χέρι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συζήτηση και ευχαριστώ για το ότι το θέμα αυτό το διατηρείτε στην Διεθνή Ατζέντα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τελείωσε η συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο θέμα το οποίο